σε λίγο. Ε, σε σχέση με την ε, γνωμοδότηση της ΟΚΕ αναφέρεται το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, των φύλων. Ε, ε δεν, ανα, δεν αναβλήθηκε και σύμφωνα με το άρθρο 137 ε, παράγραφος 2 του εσωτερικού κανονισμού το αίτημα για την ε, ε, γραμματότηση αυτή θεωρείται ως εγκριθέν. Και περνάμε στην υπόλοιπη